και δεσμεύομαι τα θέματα αυτά του Ιράν να τα θέτω και δημοσίως και ιδιωτικός. Όντως, αυτά που έχουν συμβεί είναι φοβερά και ελπίζω ότι οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν. Αυτά είναι τα γενικά. Τώρα, για να προσπαθήσω να απαντήσω στα πιο συγκεκριμένα θέματα τα οποία θέσατε, είναι σίγουρο ότι η στήριξη της ε, συμφωνίας εμπόδισε την Ευρωπαϊκή Ένωση να επικεντρωθεί σε άλλα ζητήματα. Εμείς έχουμε δεσμευτεί σε έναν ειλικρινή και ανοιχτό διάλογο με το Ιράν για όλα τα θέματα. Και διατηρούμε τη δυνατότητα για αυτόνομα περιοριστικά μέτρα, ακόμη και σε περίπτωση παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν πιστεύουμε ότι θα ήμασταν σε καλύτερη κατάσταση για να αντιμετωπιστούν αυτά τα ζητήματα χωρίς την πυρηνική συμφωνία. Και σας διαβεβαιώ, το πιστεύω ότι η GCPOA καταρχήν ε, εγκρίθηκε και από ψήφισμα του ΙΕ. Δεν ήταν δηλαδή καταρχήν κάτι το οποίο ονειρεύτηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ το ξεκίνησε. Και εμείς θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό ζήτημα για την περιφερειακή αλλά και την παγκόσμια ισορροπία. Κανείς δεν θέλει μια κούρσα για πυρηνικά όπλα και κανείς μέχρι τώρα δεν κατάφερε να βρει ειρηνικό τρόπο άλλο, ειρηνικό, έτσι για να διασφαλίσει ότι το Ιράν δεν θα αναπτύξει πυρηνικά όπλα. Κατόπιν τούτων, έχουμε πολλές ευκαιρίες. Από τον ε, Ιούνιο του 2019, το είπαμε και το ξαναείπαμε, ότι θέλουμε να τηρήσει τις δεσμεύσεις του το Ιράν και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε το στόχο και την πλήρη υλοποίηση της συμφωνίας αυτής και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να διασώσουμε αυτή τη συμφωνία για τα πυρηνικά με το Ιράν. Άλλοι λένε ότι είμαστε πολύ ήπιοι, πολύ μαλακοί με το Ιράν. Και εδώ θα ήθελα μια ειλικρινή συζήτηση. Ας δούμε τα πραγματικά ζητήματα. Είμαστε όντως πολύ μαλακοί με το Ιράν εγώ δεν νομίζω. Υπάρχουν ακόμα κυρώσεις. Πρώτον, κυρώσεις βάσει της συμφωνίας αυτής για τα πυρηνικά. Δεύτερον, κυρώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα. 83 άτομα και οντότητες όπως επίσης και απαγορεύσεις εξοπλισμού προς το Ιράν που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καταστολή, όπως επίσης και για εξοπλισμό που ελέγχεται στις τηλεπικοινωνίες. Γιατί ξέρετε ότι όταν ταράσετε την κυκλοφορία στο δίκτυο, χρειάζεστε μέσα ιδιαίτερα περίπλοκα και προηγμένα. Και τρίτον, κυρώσεις όσον αφορά τη Συρία και την τρομοκρατία. Άρα δεν νομίζω ότι είμαστε μαλακοί. Κάνουμε ό,τι πρέπει να κάνουμε. Και νομίζω ότι καταλαβαίνετε υπέροχα ότι η συμφωνία αυτή είναι σημαντική για μας, αλλά δεν μας εμποδίζει να είμαστε σκληροί εφόσον ε, χρειαστεί, όταν συμβαίνουν πράγματα όπως αυτά που είδαμε ότι συνέβησαν στο Ιράν. Και όντως, τίθεται θέμα πώς θα απαντήσουμε στην καταστολή αυτή. Η αλήθεια είναι ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν προτάσεις για να προσθεθούν ε, μέτρα ε, στον κατάλογο κυρώσεων που έχουμε. Υπάρχει το, η αναθεώρηση του καθεστώτος για τα ανθρώπινα δικαιώματα, η οποία προχωράει. Έχουμε ακόμα κυρώσεις ενισχύ, όπως σας είπα, που αφορούν 83 άτομα και οντότητες στο Ιράν. Πρόκειται για ένα δύσκολο ζήτημα. Συνεχίζουμε να δουλεύουμε πάνω σε αυτό, χρησιμοποιώντας συγχρόνως κάθε διπλωματική δυνατότητα που έχουμε. Λέμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ασφαλειά μας και από την άλλη μεριά υποστηρίζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και στο Ιράν και αλλού. Με κυρώσεις όταν χρειάζεται, με διπλωματική πίεση και επιμονή μου βάσεως ζητούμε το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτέ, κυρία Πρόεδρε, ήταν μια πολύ εντατική σύνοδος αυτή. Ήταν η πρώτη φορά ε, που ήρθα εδώ και θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για τη συνεισφορά σας, τη στήριξή σας και ξέρω ότι δεν βλέπουν όλοι με τον ίδιο τρόπο τα πράγματα από την αριστερά μέχρι τη δεξιά. Υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις, διαφορετική κατανόηση για το τι συμβαίνει σε αυτό το δύσκολο κόσμο μέσα στον οποίο καλούμεθα να ζήσουμε. Σήμερα καλύψαμε πόσα θέματα. Τέσσερα, τέσσερα δύσκολα ζητήματα. Χάρη σε εσά. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν για τη συνεισφορά σας και την στήριξή σα στα καθήκοντά μου. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι έχουν κατατεθεί έξι ψηφίσματα. Και εδώ ολοκληρώνει τη σύντηση. Αύριο θα διεξαχθεί η ψηφοφορία. Θα πρέπει να σας πω ότι το ΕΛΚ και ο πρόεδρος του μας είπε ότι θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές στις αντιπροσωπείες και τις επιτροπές του Κοινοβουλίου. Τα ονόματα των νέων μελών θα σημειωθούν στα πρακτικά της σημερινής συνεδρίασης και από σήμερα γίνονται μέλη των ε, ε, αντίστοιχων επιτροπών και αντιπροσωπιών. Ευχαριστώ πολύ. Θα συνεχίσουμε με την ημερήσια διάταξη, δηλώσει Συμβουλίου και τη Επιτροπή για τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τους ακροτηριασμούς των γεννητικών οργάνων των κοριτσιών και γυναικών. Λόγο έχει καταρχήν η κυρία του Πουράινεν εκ μέρους του Συμβουλίου. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, τα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών και η ισότητα των φίλων ήταν βασική γενική προτεραιότητα της Προεδρίας μας στα πλαίσια της αναπτύξεως και της συνεργασίας. Ακολουθήσαμε προσήγγιση βάσει των δικαιωμάτων την ανάπτυξη συμπεριλαμβανομένης και τη ε, σεξουαλική αναπαραγωγή και της υγείας. Ε, είμαστε σοβαροί όσον αφορά τι δεσμεύσει που αναλάβαμε στα πλαίσια τη Ευρωπαϊκή Συνένεση για Ανάπτυξη και του στόχου βιώσιμη ανάπτυξη. Θα να συνεργαστούμε με του εταίρου μα για να εκκριζώσουμε κάθε μορφή σεξουαλική και έμφυλη ε, βία και διάκριση συμπεριλαμβανομένων και επιβλαβών πρακτικών, όπω πιο συγκεκριμένα ο, γεν, ο γενετικό ακροτηριασμό γυναικών και κοριτσιών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη αυτή έχουν επιδείξει επιμακρών ε, ηγεσία ε, και προσπάθεια σε πολυμερέ επίπεδο για να προωθούν τα δικαιώματα των κοριτσιών και των γυναικών και την ισότητα των φύλων η πρωτοβουλία του ΕΕ προβολέ Spotlight για να εξαλειφθεί αυτή η πρακτική κατά γυναικών και κοριτσιών είναι ένα καλό παράδειγμα άνευ προηγουμένου προσπάθεια σε παγκόσμιο επίπεδο για πρόθεση ισότητα των φύλων και να δοθεί δύναμη στι γυναίκε. Και όλα αυτά να είναι προποθέσει και φορέα για την επίτευξη των στόχων βιώσιμη ανάπτυξη. Στην Αφρική, η πρωτοβουλία Spotlight ασχολείται με έμφυλη βία, σεξουαλική βία, ε, γάμο παιδιών, γενετικό ακροτηριασμό των γυναικών και πώς σχετίζονται αυτά με την πρόσβαση στην σεξουαλική και την αναπαραγωγική υγεία. Ο λόγος για τη διάσκεψη για το πληθυσμό και ανάπτυξη, συν 25, που τη φιλόξενησαν η Κένια, ε, η Δανία και αρμόδιος φορέας του ΟΗΕ στο Ναϊρόμπι ήταν μια εξαιρετικά επιτυχή συνεδρίαση και δεσμεύτηκαν, δόθηκαν χορηγίε και από ιδιωτικό φορέα και δημόσιο φορέα και ανελήφθησαν πολιτικέ υποχρεώσει και επιβεβαιώθηκε εκ νέου ότι πρέπει να γίνουν προσπάθειε για να πετύχουμε ε, μηδέν ακροτηριασμό των γυναικών μέχρι το 2030 βάσει του θεματολογίου του 2030 για την βιώσιμη ανάπτυξη. Όλα αυτά. Τα επιτέγματά μας και η ηγεσία μας είναι κάτι πραγματικό αλλά πρέπει να συνεχίσουμε να σπρώχνουμε με χρυσότου να ανταποκριθούμε στην υποχρέωσή μας να πετύχουμε το στόχο μηδέν επιβλαβείς πρακτικές κατά των γυναικών και των ε, κοριτσιών. Αξιότιμα μέλη, κυρία Πρόεδρε, τα Ηνωμένα Έθνη τις 6 Φεβρουαρίου την καθόρισαν Διεθνή ημέρα μηδενικής ανοχής για τον γενετικό κροτηριασμό των γυναικών και των κοριτσιών και εκείνη την ημέρα αποτιμά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπάθειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με αυτό. Προσβλέπουμε στη σχετική έκθεση. Επίση, επιθυμούμε διακαώς να δούμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ανανέωση της στρατηγικής δέσμευσης της Ευρωπαϊκής Ενώσης για ισότητα των φύλων που εκπνέει τέλος τρέχοντος μηνός. Αυτό ελπίζουμε να συμπεριλαμβάνει και στρατηγική Ευρωπαϊκή Ένωση, Ενώσης να τεθεί τέρμα στον ακροτηριασμό των γυναικών και κοριτσιών σε όλο τον κόσμο, άπαξ διαπαντός. Λοιπόν, κλείνοντα να υπενθυμίσω ότι δυστυχώ σημαντικό αριθμό γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση ζουν με διαβίου συνέπεια του γενετικού αυτοκρατηριασμού των γυναικών ή κινδυνεύουν. Κινδυνεύει η ζωή του από αυτό. Χωρί να αγνοήσουμε τα επιτέγματά μα, γνωρίζουμε όμω την ανάγκη να γίνουν περισσότερα στην Ευρώπη σχετικά με την εφαρμογή των εθνικών νομοθεσιών, ειδικευμένε υπηρεσίε υποστήριξη ή πολετομιακέ δράσει όσον αφορά τι πληγήσει κοινότητε. Κυρία Πρόεδρε, πιστεύω ότι συνεχίζοντας τη συνεργασία μας θα είμαστε θέση να εξασφαλίσουμε περαιτέρω επιτεύγματα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την σημαντικότατη συζήτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Η κυρία Ντάλη έχει τώρα το λόγο εκ μέρου τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που έβαλε αυτό το σημαντικό θέμα στην σημερινή μερίσια διάταξη. Και ευχαριστώ πολύ και την φιλανδική κυβέρνηση για τη δέσμευσή της σε σχέση με αυτό το θέμα και την ισότητα μεταξύ των δύο φίλων. Αυτό το θέμα είναι ένα θέμα που έχω πραγματικά στην καρδιά μου και έχω υποσχεθεί ότι θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να εξαλείψω αυτή τη μάστιγα. Αυτό το βασανιστήριο που υφίστανται τόσες πολλές γυναίκες και κορίτσια, ακόμα και σήμερα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Είναι ζωτική σημασία λοιπόν να εκθέσουμε και να καταπολεμήσουμε αυτή τη φοβερή παραβίαση ανθρωπίνων ε, δικαιωμάτων, δικαιωμάτων των γυναικών και των παιδιών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ΙΕ έχουν πρόγραμμα για την εξάλληψη κάθε μορφής βίας σε βάρος των γυναικών και των ε, κοριτσιών με 100 εκατομμύρια ευρώ και αναφέρθηκε ήδη. Αλλά σκοπός είναι να μην υπάρξει κανένα κορίτσι και καμία γυναίκα ξεχασμένη σε αυτό το δρόμο. Σε πάρα πολλές αφρικανικές ε, χώρες έχουμε βοηθήσει και έχουμε στηρίξει με αποτέλεσμα 1,5 εκατομμύριο γυναικών να έχουν τύχη φροντίδας σε σχέση με τον ακροτηριασμό αυτό. Επίσης υπάρχουν και κινήματα πολιτών σε πάνω από 3.000 κοινότητες με 8,5 εκατομμύρια άτομα που κινητοποιούνται για να υπάρξει δημόσια δήλωση για κατάληψη αυτής της πρακτικής. Ξέρουμε ότι η πρακτική αυτή υφίσταται και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μισό εκατομμύριο κορίτσια και γυναίκες έχουν υποφέρει από ακροτηριασμό γενετικών οργάνων ζώντας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όμως η προσπάθειά μας για ισότητα ε, παίζει ρόλο προκειμένου να ενημερωθεί ο κόσμος για το τι συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τον ακροτηριασμό αυτό. Σε όλες μας ε, τις χώρες θεωρείται έγκλημα ο ακροτηριασμός ε, των γυναικείων γεννητικών οργάνων και Επίση, στην νομοθεσία μας προβλέπεται τη φροντίδα για τα θύματα στα πλαίσια της οδηγίας ε, για την βοήθεια σε θύματα. Έπειτα έχουμε και την νομοθεσία μας για το άσυλο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζει να δίνει χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος ε, Δάφνη αλλά και άλλων για την καταπολέμηση της βίας που έχει να κάνει με το φύλλο συμπεριλαμβανομένου και το κρατηριασμό αυτού. Ήδη στην αρχή του 2020 θα ξεκινήσουμε ένα προπολογισμό 12,4 εκατομμυρίων ευρώ. Αξιότιμοι ευρωβουλευτέ, πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να διασφαλίσουμε ότι οι προβλέψει και εκτιμήσει για άλλα 200 εκατομμύρια θύματα μέχρι το 2030 δεν θα επαληθευτεί. Η ατζέντα για την Ευρώπη της Προέδρου Φοντερ Λάιον συμπεριλαμβάνει την πρόληψη της βίας σε βάρος των ε, γυναικών και έχει θέσει αυτό το θέμα στην, ε, στον πυρήνα, στην καρδιά της δράσης μας για την επόμενη πενταετία. Και είμαι σίγουρη ότι μπορώ να βασιστώ στη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για αυτό το θέμα. Η επόμενη στρατηγική για την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων που θα εγκρίνουμε το 2020 θα συμπεριλαμβάνει και τη βία σε βάρος των γυναικών και θα προβλέπει διάφορα μέτρα και κατά του ακροτηριασμού γυναικείων γενετικών οργάνων. Θέλουμε να δράσουμε σε πολλούς άξονες συγχρόνως, να δούμε το θέμα από διαφορετικά πρίσματα και οπτικές γωνίες, και να το συμπεριλάβουμε σε διάφορα χαρτοφυλάκια. Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε στις, στους πέντε τομείς προτεραιότητας που αναφέρονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής για το 2030 προκειμένου να καταργηθεί η πρακτική αυτή της, του ακροτηριασμού ε, γεννητικών γυναικείων οργάνων. Θέλουμε να υπάρξουν και κοινωνικές αλλαγές, προστασία, δίωξη και η καταπολέμηση της πρακτικής αυτής παγκοσμίω. Τα δικαιώματα των γυναικών βρίσκονται στην καρδιά της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμπεριλαμβάνει και την καταπολέμηση της πρακτικής αυτής. Πρέπει να συνεργαστούμε με τους διεθνείς εταίρους μας ανά τον κόσμο για να στηρίξουμε την η υλοποίηση των στόχων βιώσιμη ανάπτυξη που συμπεριλαμβάνει και την καταπολέμηση τη βία σε βάρο των γυναικών. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σημαντικό ρόλο να παίξει με τα δίκτυα που έχει ανά τον κόσμο. Συγχρόνω αναγνωρίζουμε ότι η πρακτική αυτή είναι ένα ευαίσθητο θέμα για να το αντιμετωπίσουμε. Γιατί έχει διάφορες πτυχές και ανθρώπινα δικαιώματα και δικαιώματα ε, γυναικών και σωματική ακερότητα και βία, αλλά και το δικαίωμα στην υγεία. Γι' αυτό είναι σημαντικό να συνεργαστούμε με επιζήσαντες από την πρακτική αυτή ή με τις κοινότητες οι οποίες ε, εφαρμόζουν αυτή την πρακτική, να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις ούτε προκαταλήψεις. Πρέπει να αποφύγουμε επίσης το στιγματισμό, το ρατσισμό και την ξενοφοβία. Πάση θυσία. Πρέπει να προωθήσουμε τη συνεργασία και το διάλογο. Πέρα από τη χρηματοδότηση και την νομοθεσία, πρέπει να συμπεριλάβουμε στη δράση μας και όλους τους ενδιαφερόμενους σε όλα τα επίπεδα πολιτικό διάλογο με τις εθνικές κυβερνήσεις, στήριξη στους επαγγελματίες του κλάδου της υγείας, επικεφαλής κοινοτήτων, οικογένειες, προκειμένου να καταργηθεί μια για πάντα η πρακτική αυτή. Προσβλέπω στις δικές σας απόψεις και προσβλέπω επίσης τη συνεργασία μαζί σας για να πετύχουμε αυτό τον τόσο σημαντικό στόχο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Εκ μέρους του ΑΕΛΚ έχει το λόγο η κυρία Φιτζέραλτ. Ευχαριστώ. Καλωσορίζω ήδη αυτά που υπόθηκαν σήμερα από τους εκπροσώπου του Συμβουλίου και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το οικοτηριασμό γενετικός των γυναικών είναι ένας ορισμός που αφορά τον πολιτισμό, την παράδοση και είναι, θεωρείται και ιατρική ε, παρέμβαση. Αλλά στα αρχικά δεν βλέπουμε καμία από τι τρει το FGM. Είναι μια επίθεση. Βία, βία κατά των γυναικών ουσιαστικά και βία κατά των γυναικών που καταλήγει σε θεμελιώδεις τραυματισμούς που διαρκούν μια ζωή. Τραύματα που βλάπτουν την ε, γυναίκα και αλλάζουν το νόημα του να είναι ένας άνθρωπος γυναίκα. Από το 2018, τον Οκτώβριο 2018, υπολογίστηκε ότι 2 εκατομμύρια γυναίκες και κορίτσια έχουν περάσει αυτόν τον ακροτηριασμό σε 30 χώρες. Και αυτό είναι απλώς μια εκτίμηση, να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα με πολλές ε, περιπτώσεις που δεν αναφέρονται, δεν καταγγέλλονται. Όταν σκέφτονται αυτόν τον κοτιδιασμό, οι περισσότεροι σκέφτονται την Αφρικανική Ήπειρο, την Γουινέα που 45% ε, κοριτσιών κάτω από 14 ετών. Όπω η Αιθιοπία, 65% των γυναικών έχουν περάσει αυτόν τον ακροτηριασμό. Αλλά η πραγματικότητα ποια είναι. Συμβαίνει και σε χώρε όλο τον κόσμο, σε μέρη όπω είναι η Ινδονησία, όπω είναι η Μαλαισία και ούτω καθεξής. Τι θα μπορούσαμε να πούμε αν αυτή ήταν η μητέρα μα, η αδελφή μα, η γυναίκα μα, τα ξαδέλφια μα θα ήμασταν τόσο καθησυχασμένοι όπω είμαστε μερικέ φορέ. Θα ήμασταν εξωφρενών και θα πρέπει να είμαστε οι φωνέ αυτών των γυναικών που δεν μπορούν να μιλήσουν για τον εαυτό του. Θέλουμε να προσπαθήσουμε ώστε η διάσκεψη, η σύμβαση τη Κωνσταντινούπολη εφαρμοστεί. Είναι βία κατά των γυναικών αυτό ο ακροτηριασμό και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάθε θέσιμο πόρο για να κρυζώσουμε αυτό το φαινόμενο. Πώ το καταφέρνουμε αυτό, θα πρέπει να γίνει σοβαρή ύψιστη προτεραιότητα, να γίνει προσπάθεια συγκεκριμένη αυτό το θέμα. Χρειάζεται πολιτική ηγεσία, τους πολιτικούς ηγέτες όλο τον κόσμο, γυναίκες και άντρες. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε σε παγκόσμιο πολυεπίπεδο σύστημα με πολλούς ενδιαφερόμενους ΜΚΟ, κοινότητες, οικογένειες. Πρέπει να συνεργαστούν όλοι μαζί. Η UNICEF συνεπέρανε ότι διεξήγαγε από τη διεξαγωγή των ερευνών τη ότι οι περισσότερε γυναίκε στα κορίτσια, στι περισσότερε ε, χώρες πιστεύουν ότι πρέπει τέρμα. Χρειαζόμαστε διάφορους οι οποίοι μπαίνουν στην πρώτη γραμμή. οι που και διάφορες γυναίκες που εργάζονται για να εκριζώσουν αυτόν τον ακροτηριασμό. Η βία κατά των γυναικών είναι ένα έγκλημα, είναι ένα έγκλημα ακροτηριασμό αυτό και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε από την πλευρά μας να το σταματήσουμε αυτό το φαινόμενο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Εκ μέρου των ε, σοσιαλδημοκρατών έχει το λόγο η κυρία Νόχλε. Δυστυχώς το σώμα των γυναικών είναι ένα πεδίο μάχης σε κάθε πολιτισμό, σε κάθε θρησκεία, σε κάθε ήπειρο και ε, σε όλες τις ιστορικές περιόδους. Και είναι πάντοτε το γυναικείο σώμα αυτό το οποίο ε, γίνεται θύμα επίθεσης. Πώς μπορούμε να το εξηγήσουμε. Μπορούμε να θυμηθούμε τι έγινε στην Κίνα. Ήταν το γυναικείο σώμα, ήταν τα πόδια των γυναικών που το έδαιναν έτσι, που ήταν μια ουσιαστική αναπηρία. Δεν ήταν ποτέ οι άντρε που του έδαιναν τα πόδια. Ήταν ε, οι γυναίκε που έπεφταν ε, επίση ε, θύμα του κορσέ. Και αυτό που γίνεται στο παρόν τώρα, η αναπηρία των γενετικών οργάνων που στερεί από τις γυναίκες την σεξουαλική τους ελευθερία, τους δημιουργεί πόνους ισοβίας. Ε, και πολλές φορές ράβουν και τον κόλπο στις γυναίκες, όχι στους άνδρες τα γενετικά όργανα. Επίσης, ο πολιτισμός, η αντίληψη της παρθενίας ε, και απαντάται και στην Ευρώπη. Και πάντοτε το θέμα είναι το εξής. Ο έλεγχος των ανδρών στα γυναικεία σώματα ε, πρόκειται για μια παρέμβαση στο γυναικείο σώμα και πρόκειται για μια προσπάθεια να προκαλέσει κανείς πόνο στο γυναικείο σώμα. Ευχαριστούμε πολύ. Εκ μέρους του Ρινιού η κυρία Τολερέ έχει το λόγο. Σήμερα 500.000 γυναίκες στην Ευρώπη και 2 εκατομμύρια στον κόσμο είναι θύματα αυτού του γενετικού κροτηριασμού των γυναικών. Η ζωή τους, η ιδιωτική, η ζωή τους, η γυναικεία επηρεάζεται και μόνος τους πρέπει να υποστούν τις συνέπειες. Θα πρέπει να εκριζωθεί αυτή η μάστιγα και για αυτό το σκοπό να εθετήσουμε μια κοινή προσπάθεια ρεαλιστική, καταρχάς εξασφαλίζοντας τη συλλογή και την διάδοση των στοιχείων. Χρειαζόμαστε στοιχεία που είναι ακριβή, συγκρίσιμα δεδομένα και να έχουμε αδιαφυσβήτητα αριθματικά στοιχεία για να προσμετρήσουμε την εξέλιξη και στην Ευρώπη. Χρειαζόμαστε συνεργασία μεγάλη, ευρεία, να εφαρμόσουμε προληπτικά μέτρα που θα κινητοποιήσουν όλους τους φορείς συμπεριλαμβανομένων και των πληττωμένων κοινοτήτων. Επίσης, χρειαζόμαστε μέτρα υποστήριξης, προστασίας και νομικής κάλυψης όλων των ατόμων που πλήττονται. Κυρία Επίτροπε, σήμερα έχουμε όλα τα μέσα στα χέρια μας για να διευθετήσουμε το πρόβλημα. Χαιρετίζω τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μην λησμονήσει την στρατηγική που θα εφαρμόσει την ισότητα και καταπολεμά το πρόβλημα του γενετικού ακροτηριασμού των γυναικών. Έχουμε και την ε, σύμβαση της Κωνσταντινούπολης που αναφέρεται σε αυτό το φαινόμενο που δεν επικυρώθηκε από 7 κράτη-μέλη ακόμα. Εμείς οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να είμαστε η φωνή αυτών των γυναικών και της οργής τους. Με τον παρόντα αριθμό 68 εκατομμύρια κορίτσια θα εκτεθούν ανάμεσα στο 2015 και το 2030 στο γενετικό ακροτηριασμό των γυναικών αν δεν κάνουμε τίποτα. Είναι απαράδεκτο, δεν πρέπει να αφήσουμε να γίνει. Έχετε κάθε υποστήριξη από εμά για να εφαρμόσετε αυτή τη στρατηγική. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Επόμενη ομιλήτρια είναι η κυρία Χέρτσπεργκελ οι περισσότερες παρεμβάσεις αυτές έχουν σαν στόχο να ακροτηριάσουν τα γυναικεία σώματα για μη ιατρικούς λόγους και πρόκειται για μια κατάφορη παραβίαση των δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών. Αυτή η πρακτική παραβιάζει επίσης το δικαίωμά τους στην ε, σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία καθώς και τη σωματική τους ακαιρεότητα. Οι ακροτηριασμοί είναι καθολικό φαινόμενο το οποίο πλήττει τόσο τις αφρικανικές χώρες όσο και τις χώρες Αγγής Ανατολής, της ε, Ευρώπης επίσης. Ε, στην η Γερμανία 20.000 γυναίκες και 4.000 νερά κορίτσια έχουν ακροτηριαστεί. Ε, τα θύματα τα οποία έχουν επιζήσει στην Ευρώπη είναι περίπου 5.000. Οι, γενετήσιοι ακροτηριασμοί ε, βασίζονται σε σφαλμένες ε, θρησκευτικές πεπιθήσεις. Παρά την ε, νομοθεσία η οποία ισχύει σε πολλές χώρες της Αφρικής υπάρχουν θηλαίκοι αντίστασης. υπάρχουν, γίνονται εξαρτίες ευαισθητοποίησης προκειμένου να εξαλειφθεί αυτό το φαινόμενο. Πρόκειται για παραχημένες παραδόσεις οι οποίες ε, αφομοιώθηκαν ε, στην ε, Ισλαμική θρησκεία, εσφαλμένα. Ούτε στο Κοράνι, ούτε στη Βίβλο, ούτε στη Τώρα δεν, δεν διατυπώνεται η απέτηση να ακροτηριάζονται οι γυναίκες. Πρόκειται για πρακτικές που γίνονται με τη συμμετοχή νέων ανθρώπων με τη συμμετοχή συγγνώμη των διαφόρων θα πρέπει να σπάσουμε τα ταμπού μέσω της πρόληψης και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να, να προσανατολίσουμε ε, τους ανθρώπους αυτούς προς άλλες δραστηριότητες, ούτε ώστε οι κοινότητες αυτές ε, να μην στιγματίζονται μεν, αλλά να προχωρήσουν στην κατάργηση αυτών των πρακτικών. Θα πρέπει να προστατευτεί η σωματική ακαιρεότητα των γυναικών και των κοριτσιών σε ένα πνεύμα αλληλοσεβασμού, ούτως ώστε να ε, μπορέσουμε να εξαλείψουμε ριζικά το φαινόμενο. Παλεύουμε για την, απάλυψη, για την κατάργηση ενός φαινομένου βίας, το οποίο πλήττει την υγεία των γυναικών και των κοριτσιών. Παρακαλώ να τηρείτε το χρόνο αγόρευσης. Η επόμενη ομιλήτρια είναι η κυρία Άντερσον. Μιλούμε εδώ για την στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση μιας πρακτικής ακροτηριασμού των γυναικών η οποία συνιστά μια πράξη περιφρόνησης των γυναικών. Ε, ακούσαμε από τους ε, προλαλήσαντες ε, ότι θα πρέπει να καταπολεμωθούν αυτή η πρακτική από ορισμένου συναδέλφου. Αλλά πρόκειται για μεγάλη υποκρισία, γιατί ακριβώς οι συνάδελφοι αυτοί κατέθεσαν, ε, ε, ε, μάλλον αρνήθηκαν την προσπάθεια μιας, ενός ψηφίματος το οποίο θα καταδίκαζε αυτές τις πρακτικές. Για ποιο λόγο γιατί το πεπρωμένο αυτών των γυναικών τους είναι απολύτως αδιάφορο. Για εκείνους είναι πολύ πιο σημαντικό να καταψηφίσουν αυτό το ψήφισμα το οποίο προέρχεται ε, από μένα που είμαι άτομο νον γκράτα για αυτούς τους ανθρώπους. Η δική μου τροπολογία στο ψήφισμα ε, είχε σαν σκοπό να τονίσει την αποφασιστικότητα με την οποία καταδικάζουμε αυτή την αποτρόπαια πρακτική. Όμως ε, μέσω της απόρριψης αυτής της τροπολογίας ε, ο γυναικείος ακροτηριασμός απλώς αναφέρεται με τη μορφή μιας υποσημείωσης. Σε ποιον πουλάτε τέτοια ψέματα ότι θέλετε να καταπολεμήσετε αυτές τις πρακτικές του γυναικείου ακροτηριασμού. Ε, σήμερα οι βουλευτές ε, Παλόπ, Μαγκίνες, ε, Περέρα, Τζόνς και και εκείνοι καταψήφισαν αυτή την τροπολογία. Υποκρίνεστε ότι σας αφορούν, ότι σας φύγουν αυτά τα θέματα αλλά με τον τρόπο αυτό δείχνετε ε, την περιφρόνησή σας προς την εισηγήτρια. Η κυρία Κάνκο εκ μέρους των Ευρωπαίων Συντηρητικών. Έχει να κάνει με κάθε φάση της ζωής σας ο κρατηριασμός αυτός. Επηρεάζει τον άνθρωπο σαν άνθρωπο, την εμπιστοσύνη του παιδιού. Πώς ε, αισθάνεσαι πώς νιώθεις όταν ε, περιμένεις παιδί, όταν γεννάς, πώς αγαπάς τους ενήλικες και πώς αγαπάς τον εαυτό σου και μεταχειρίζεσαι τον εαυτό σου. Είναι μία παραβίαση. Καταστρέφει το σώμα σου, το μυαλό σου. Είσαι χωρίς να μπορείς να κάνεις τίποτα ανυπεράσπιστος όταν είσαι παιδί. Απλώς προσπαθείς να επιβιώσεις. Δεν θέλεις, αλλά πρέπει για να μην ξεχάσεις ποτέ ότι η αξία σου είναι η ίδια αξία όπως και οποιοδήποτε άλλου. Και εγώ αυτό τον αγώνα δίνω καθημερινά. 200 εκατομμύρια γυναίκες και παιδιά ανά τον κόσμο και 500.000 εδώ στην Ευρώπη, τα καθημερινά θύματα. Η αλλαγή πάει πολύ αργά και είναι πολύ μικρή. Επιγόντως χρειαζόμαστε στρατηγικές και ένα πρόγραμμα δράσης που να έχει πραγματικά αντίκτυπο. Εγώ συγκινήθηκα και εμπνεύστηκα πάρα πολύ από τους restorers, αυτού που βοηθούν στην αποκατάσταση των ε, νέων ε, γυναικών που έχουν υποστεί τέτοιον ακροτηριασμό. Πρέπει να ξέρουμε ότι όποιες επιλογές και αν κάνουμε, υπάρχει κάπου ένα κορίτσι που το όνειρά του και η ζωή του εξαρτώνται από εμά. Πρέπει πρώτα απ' όλα λοιπόν να τους δούμε, ε, να, να τα δούμε αυτά τα παιδιά, να τα ακούσουμε και να τα βοηθήσουμε να χρησιμοποιήσουν τις δυνάμεις τους και να ζήσουν ένα ελεύθερο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Τώρα η κυρία Ροντρίγκε Πάλοπ έχει το λόγο εκ μέρου τη ΓΚΟΕ, παρακαλώ. Ο ακροτηριασμό των γυναικών είναι μια ματσιστική πρακτική και παραβίαση των δικαιωμάτων των γυναικών και των αναπαραγωγικών τους. Το πρόβλημα είναι ότι πολλοί χρησιμοποιούν ε, τη συζήτηση για την πρακτική αυτή για να επιβραβεύσουν το λόγο της Ευρώπης υπέρ του ρατσισμού. Ο ακροτηριασμός υπάρχει και στη Μέση Ανατολή και στη Λατινική Αμερική, δεν είναι μόνο στην Ασία και ακόμα και στην Ευρώπη και στις Ηνωμένε Πολιτείε προκειμένου να θεραπευθούν λέει, κάποιες ασθένειες όπως ήταν η γυναική αστερία είναι θρησκευτική πρακτική, αλλά όχι μόνο των μουσουλμάνων και οι κόπτες χριστιανοί και κάποιοι άλλοι επίσης ούτε το εφαρμόζουν. Μην ξεγελιόμαστε. Διακόπτη πρόεδρος, κοιτάξτε, μιλάτε λίγο πιο αργά γιατί είναι αδύνατο να μεταφραστείτε. Δεν μπορεί να σας παρακολουθήσουν οι διερμηνείς η δεξιά και άκρα δεξιά δεν νοιάζεται ούτε για τα κορίτσια ούτε για τις γυναίκες και τον ακροτηρισμό. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι η σταυροφορία για το δικό τους τρόπο να αντιλαμβάνονται το χριστιανισμό. Γι' αυτό συνεχίζουν την πρακτική και δεν θέλουν την σύμβαση της Κωνσταντινούπολης που είναι ο μόνος τρόπος που έχουμε για να σταματήσουμε με αυτή την πρακτική. Η κυρία Γουόλς έχει το λόγο. Από το ΕΛΚ. Συνάδελφοι, με απογοητεύει η προγραμματίστηκε στο τέλο τη ημέρα αυτή η συζήτηση και δεν δόθηκε η πλατφόρμα που αξίζει με περισσότερη παρουσία ανδρών και γυναικών με τα 28 κράτη-μέλη να συμμετέχουν ενεργά. Είναι σαφέστατο ότι ο γενετικό ακροτηριασμό των γυναικών δεν έχει ωφελήσει τα 200 εκατομμύρια γυναίκε και κορίτσια που το έκαναν αυτό. Του το έκαναν αυτό και να πάμε πιο κοντά στην πατρίδα μα δεν θα ωφελήσει τι 180.000 κορίτσια και γυναίκες που κινδυνεύουν να υποστούν αυτόν τον ακροτηριασμό εδώ στην Ευρώπη. Γίνεται για να ελέγξουν τα κορίτσια και τις γυναίκες, τα σώματά τους, γίνεται για να ελέγξουν τις ζωέ που ζουν και τις ζωέ που τους αξίζει να ζήσουν και γίνεται με ψεύδο ιδεολογία, σύμφωνα την οποία ότι μια, ένα κορίτσι θα μπορούσε να ωφεληθεί από αυτόν τον ακροτηριασμό. Εμείς Όλοι εμεί πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι οι επιβλαβεί πρακτικέ όπω ο γενετικό εκοτιασμό των γενετικών κοριτσιών δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί απομονωμένα. Θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ολιστικά, ε, σφαιρικά, για να σταματήσει κάθε μορφή βία. Και θέλουμε μια στατική τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω που θα απαγορεύει ε, αυτό τον ακροτηριασμό για να προστατεύσουμε μελλοντικέ γενιέ γυναικών και κοριτσιών. Πολιτικά μέτρα πρέπει να εστιάζονται κοινοτήτων, παραδοσιακών ηγετών θρησκειών, ανδρών γυναικών, να του παρουσιάσουμε σαν φορεί αλλαγή αυτή η αναγνώριση είναι ένα κρίσιμο βήμα, δεν αρκεί όμως. Εμείς, και λέω εμείς όλοι μαζί, πρέπει να αναποκριθούμε στις υποχρεώσει που αναλάβουμε και να αναγνωρίσουμε ότι έχουμε πραγματικές ευθύνες εντός της παγκόσμιας κοινότητας και να θέσουμε τέρμα σε αυτό το κινητικό κριτισμό των κοινωνικών. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Ward έχει το λόγο για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, εκτιμάται ότι πάνω από 200 εκατομμύρια κορίτσια και γυναίκες που ζουν σήμερα έχουν υποστεί γενετικό ακροτηριασμό σε χώρες όπου πρακτική συμβαίνει και αυτό συμπεριλαμβάνει και κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Έτσι δε περαιτέρω, εκτιμάται ότι 3 εκατομμύρια κορίτσια κινδυνεύουν να υποστούν αυτόν τον ακροτηριασμό κάθε χρόνο. Αυτός ο ακροτηριασμός είναι μια μορφή βίας κατά γυναικών και κοριτσιών. Δεν είναι πολιτιστική πολιτική που μπορούμε να την υπερασπιστούμε, αλλά είναι πατριαρχική εκδήλωση. Πρέπει να τεθεί τέρμα στον ακροτηριασμό, πρέπει να συνεργαστούμε με όλου του τομεί κοινωνία, να εκπαιδεύσουμε τι κοινότητε και του ε, κοινότητε, να δώσουμε τη δύναμη στα κορίτσια και τι γυναίκε να αποκτήσουν έλεγχο των, των κορμιών του και να πείσουμε και του άντρε να κινηθούν κατά αυτού. Ε, ε, βρήκα ε, κάποια κορίτσια από την Κένια σήμερα που είναι υποψήφιοι το βραβείο Ζαχάροφ για την ελευθερία της σκέψης. Αυτά τα κορίτσια δημιούργησαν μια εφαρμογή, ICAT λέγεται, που βάζει τη δύναμη στα χέρια εκείνων που κινδυνεύουν και μπορούν να, μπορούν να, να δώσουν σήμα σε οποιοδήποτε κοντινή αρχή που να βοηθήσει. Αυτά τα κορίτσια και άλλα παρόμοια όντα μπορούν να βοηθήσουν τους γειτονέ τους. Ευχαριστώ πολύ. Συνάδελφε Μπιλμπάου Μπαραντίκα έχετε το λόγο εκ μέρου του Ρινιού. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο γυναικείος ακροτηριασμός συνεχίζει να ισχύει και απειλεί εκατομμύρια γυναίκε τόσο στην Αφρική όσο και στην Ευρώπη. Είναι παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είναι η άρνηση της ισότητας μεταξύ των δύο φύλων και μια επίθεση κατά της παιδικής ηλικίας. Ε, ξεκινάμε, επιφελείται μάλλον από ένα κενό που είναι στην εκπαίδευση, στην πρόληψη. Η Ευρώπη λοιπόν πρέπει να είναι στην πρώτη γραμμή για να σταματήσει ο εφιάλτης αυτός ε, του καταλόγου απειλών σε βάρος των γυναικών. Πάρα πολλά εργαστήρια σε περιφερειακό επίπεδο και σε εθνικό ε, προσπαθούν να τους βοηθήσουνε και υπάρχουν πρωτόκολλα σε διάφορες περιοχέ ε, του κόσμου, όπως στη χώρα των Βάσκων, που βασίζονται στα σχολεία και στα κέντρα υγείας με μία συνολική στρατηγική. Εκπαίδευση λοιπόν, υγεία, κοινωνικές υπηρεσίες, δικαιοσύνη. Με συντονισμό συνεργάζονται. Ένα δίκτυο προστατεύει τις οικογένειες. Επιμορφώνει ε, παιδιά, μεγάλους, προλαμβάνει, θεραπεύει και προβλέπονται και μέτρα συνεργασίας εκτός Ευρώπης ώστε να αποφελούμεστε από τις γνώσεις που έχουμε. Ας ε, εμπνευστεί και η Επιτροπή και ας αποφεληθεί από αυτή την εμπειρία. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Αντεσούτερ, από τους Πρασίνους. Κύριε Κυρία Επίτροπε, κύριε Πρόεδρε, ο γυναικείος ακροτηριασμός είναι μια από τις πιο ακραίες πρακτικές προκειμένου να ελέγχονται τα σώματα των γυναικών και των κοριτσιών ως ε, γυναικολόγος ο οποίος ε, προσπίζεται τα ε, ανθρώπινα δικαιώματα, καταδικάζω ρητά αυτές τις πρακτικές που προκαλούν τρομερό πόνο. Ακούσαμε τους αριθμούς 200 εκατομμύρια γυναίκες, 5.000 στην Ευρώπη, κορίτσια τα οποία κινδυνεύουν ε, σε όλες τις χώρες μεταξύ όλων των κοινωνικών ε, πληθυσμιακών ομάδων. Θα πρέπει οι πρακτικές αυτές να τερματιστεί. Πρέπει τόσο οι γυναίκες όσο και οι άνδρες να υψώσουν το ανάστημά τους και να καταδικάσουν αυτές τις πρακτικές. Οι πολιτικοί από όλες πολιτικές ομάδες θα πρέπει να τις καταδικάζουν χωρίς να πέφτουν σε ρητορίε μίσους. Η Ευρώπη θα πρέπει να έχει μια, έναν ηγετικό ρόλο προκειμένου να τερματιστεί αυτή η πρακτική σε ολόκληρο τον κόσμο και γι' αυτό θα ήθελα ήθελα να κάνω μια έκκληση ε, προκειμένου να τερματιστεί ε, τώρα αυτή η πρακτική. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ε, το λόγο έχει η κυρία Ζωρό. Ε, είμαι σοκαρισμένη από τις πολυάριθμες ε, περιπτώσεις γυναικών που υπέστησαν αυτόν τον ακροτηριασμό που ε, είναι μια ακραία πρακτική βίας κατά των γυναικών. Ο ακροτηριασμός σημαίνει ότι κόβεται η κλειδωρίδα αυτών των γυναικών. Πρόκειται για εργαλεία βασινισμού που πλήττουν την εξωπρέπεια των γυναικών η, η αλήθεια είναι ότι στις χώρες μας εφαρμόζονται αυτές οι βάρβαρες πρακτικές. 20% ε, κοριτσιών που προέρχονται από χώρες όπου εφαρμόζονται αυτές οι πρακτικές είναι ένας πληθυσμός που βρίσκεται σε κίνδυνο στις ευρωπαϊκές χώρες. Πρόκειται για αριθμούς απαράδεκτους. Ε, τι είδου κοινωνίε είναι αυτή ε, όπου τόσα κορίτσια ζουν με αυτό το φόβο ότι μπορεί να ακροτηριαστούν. Η πολιτική μου ομάδα πρότεινε μία τροπολογία για αυτές τις ε, βαρβαρικές πράξεις. Ε, καταδικάσαμε αυτές τις πρακτικές και προτείναμε κάποια μέτρα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν αλλά δυστυχώ απορρίφθηκαν. Πάρα πολλοί ευρωβουλευτέ τι καταψήφισαν. Η πρακτική αυτή βασίζεται σε κάποιες πολιτισμικές ε, ε, ε, παραδόσεις που όμως δεν είναι οι δικές μας παραδόσεις. Η γαλλική νομοθεσία δεν είναι αρκετά ισχυρή ούτε ώστε να θέσει ένα τέρμα σε αυτές τις πρακτικές. Θα πρέπει λοιπόν στις χώρες αυτές να διώκονται άμεσα αυτές οι πρακτικές θα πρέπει να δώσουμε ένα τέλος σε αυτή την έλλειψη θάρρος, σε αυτή την ανοχή της ε, βαρβαρότητας. Ε, η Μαρία Κιουρί ε, ήταν Γαλλίδα. Μέλημά μας είναι να προστατεύσουμε την Ευρώπη λίκνο της, του σεβασμού της ελευθερίας για όλους. Σας ευχαριστώ. Κυρία Στέγκρουτ, ECR. Ο γυναικείος ακροτηριασμός ε, λαμβάνει χώρα στην Αφρική αλλά και στην Αγγλική Ανατολή και στην Ευρώπη ακόμα, γιατί γνωρίζουμε ότι στη Γαλλία ε, πλήττονται 60.000 γυναίκες, αλλά και στην Σουηδία υπάρχουν περίπου 15.000 γυναίκες που έπεσαν θύματα αυτής της πρακτικής και το μερίδιο των γυναικών αυτών που πλήττονται σε ολόκληρη την Ευρώπη είναι πραγματικά ε, τόσο μεγάλο που μας ανησυχεί. Πουθενά μια τέτοια πρακτική δεν έχει το, τη θέση της στην Ευρώπη. Και θεωρώ ότι η αστυνομία αλλά και οι υπηρεσίε υγείας θα πρέπει να ευαισθητοποιηθούν ούτως ώστε να τερματιστεί αυτή η πρακτική. Ε, δεν είναι δυνατό να καταργήσουμε αυτή την πρακτική σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά στην Ευρώπη πραγματικά φέρουμε την ευθύνη να το πράξουμε μέσω ενημερωτικών εκστρατιών και μέσω μιας ενισχυμένης ε, ε, συμμετοχής των κοινοτήτων, ούτω ώστε η προσπάθεια αυτή να γίνει μια πολιτική προτεραιότητα, γιατί τέτοιες πρακτικές θα πρέπει να, να πάψουν άμεσα. Επόμενη ομιλήτρια είναι η κυρία Περέιρα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ο γενετικό εκοτιασμό των γυναικών αναμφισβήτητα είναι μια ορφή βία κατά των γυναικών που ασκείται κατά τη διάρκεια τη παιδική ηλικία και δημιουργεί φυσικέ βλάβε και όσον αφορά τη σεξουαλική και συναισθηματική υγεία που διαρκεί όλη τη ζωή. Είναι μια πρακτική που πλήττει πάνω απ' όλα του πιο αδυνάμου. Οι νέε γυναίκε μέχρι 15 ετών είναι θύματα των φτωχών τάξεων θα πρέπει να γίνει ποινικό αδίκημα αυτή η πρακτική. Θα πρέπει να προληφθεί μέσω ευαισθητοποίηση όσον αφορά τι κοινότητε τι οποίε λαμβάνει η χώρα το φαινόμενο και να εκπαιδεύσουμε τι μελλοντικέ γενιέ των γυναικών. Κατά την άποψή μα, η, καταπολέμηση και κρίζωση της του γενετικού ακροτηριασμού των γυναικών συνδέεται άρρηκτα με μια ενίσχυση των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων των γυναικών και, τη μάχη για την δυνατότητα πρόσβασης στην παιδεία και στην σεξουαλική εκπαίδευση. Είναι μια μάχη για να βελτιωθεί η υγεία των παιδιών. Το φαινόμενο του γενετικού ακροτηριασμού θα ξεπεραστεί μόνο αν σημειωθεί η πρόοδο σημαντική για τι γυναίκε Γι' αυτό πολεμάμε. Σα αλέχω για το ΕΛ έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Τα νούμερα της μάστιγας αυτής είναι φοβερά και αντικατοπτρίζουν μόνο μερικό την πραγματικότητα και ατελώς. Η πραγματικότητα που βλέπουμε εμείς πέρα από τον γενετικό ακροτηριασμό βλέπουμε ότι υπάρχουν και πολλές άλλες πρακτικές που ονομάζονται πολιτισμικές και έχουν σαν αποτέλεσμα γυναίκες και τα κορίτσια να είναι τα θύματα. Η πολυγαμία, η καταναγκαστική γάμη, η μεταξύ συγγενών, η επιλεκτική άμβλωση, οι ρογμές στο σώμα των κοριτσιών, απαγόρευση των κοριτσιών να συμμετέχουν σε κάποιες ε, εκπαιδευτικέ δραστηριότητε όπως είναι ο αθλητισμό ε, ή άλλε και το ντύσιμο που του επιβάλλεται. Όλες αυτές οι πρακτικές καταδεικνύουν ότι το λεγόμενο πολυπολιτισμικό μοντέλο, το οποίο έχει υπερτιμηθεί δίχω άλλο, βασίζεται σε ένα μεγάλο βαθμό στην παραβίαση των δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών. Οφείλουμε λοιπόν να προλαμβάνουμε και να διορθώνουμε και να δώσουμε σημασία στο σχολείο, στις υπηρεσίες υγείας και τις κοινωνικές υπηρεσίες. Οφείλουμε οι πρακτικές αυτές να μην μένουν ατιμωρητοί. Χρειάζεται λοιπόν γρήγορα να ακυρώσουμε τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και όλες οι χώρες μέλη να φροντίζουν να ισχύει η δίωξη έξω εδαφικά όταν υπάρχει τέτοιο έγκλημα. Και έχουμε και την υποχρέωση να βοηθούμε τα θύματα. Και με τις διαδικασίες ασύλου όσες βρίσκονται στις επικράτειές μας να τυχαίνουν βοήθειας από μας βάσει των πρωτοκόλων που προβλέπονται για περιπτώσεις βίας σε βάρος των γυναικών. Το να κοιτάμε προς την άλλη μεριά, το να ανεχόμαστε κάποια πράγματα, δεν σημαίνει ότι σεβόμαστε άλλες πολιτισμικές συνήθειες, όχι, αλλά αγνοούμε τον νόμο, αγνοούμε την ισότητα και πλήττουμε την αξιοπρέπεια των γυναικών. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Jones, εκ μέρους των Σοσιαλδημοκρατών τώρα παρακαλώ. Θα σας ευχαριστήσω για το χρόνο, κυρία Υπουργέ και κυρία Επίτροπε. Γνωρίζουμε ότι ο γενετικός εγκοτεριασμός είναι παγκόσμιο φαινόμενο, συμβαίνει σε κάθε χώρα του κόσμου, συμβαίνει σε κορίτσια. Ξέρουμε ότι τα κορίτσια που ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν υποστεί αυτόν τον ακροτηριασμό, περίπου 2.000 στην Ουαλία, τη χώρα που εκπροσωπώ και είναι πολύ μικρή. Οι διώξει είναι πολύ ελάχιστε, πολύ λίγε. Στον Ηνωμένο Βασίλειο ε, διώχθησαν ε, περιπτώσει 30 ε, χρόνια μετά που κηρύχθηκε παράνομη πρακτική. Δίνεται ελάχιστη προσοχή στι σοβαρέ συνέπειε που έχει για τα κορίτσια και τι γυναίκε. Πέρσι η Ουαλή άνοιξε την πρώτη κλινική τη με συγκεκριμένο ιατρική υποστήριξη και ηθική υποστήριξη για επιβιώσαντε του ακροτηριασμού. Ειδικέ υπηρεσίε όπω αυτέ είναι ζωτική σημασία. Όμω αυτέ οι υπηρεσίε που κινδυνεύουν, αυτέ κινδυνεύουν περισσότερο μετά τον Brexit λόγω περικοπή απώλεια των χρημάτων τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Χρειάζεται να βοηθήσουμε τι γυναίκε, ε, να τι στηρίξουμε και τα κορίτσια και οι υπεύθυνοι να πληρώνουν. Έχουμε τη σύμβαση τη Συμβάση τη Κωνσταντινούπολη και το ΣΥΝΤΟ. Είναι δύο ισχυρά εργαλεία για την καταπολέμηση τη βία κατά των κοριτσιών και των γυναικών, συμπεριλαμβανομένου και του γενετικού ακροτηριασμού, αλλά δεν εφαρμόζονται στον Ηνωμένο Βασίλειο. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε νομοθετικά εργαλεία όπω αυτά σε μια ολιστική προσέγγιση και ανέφερα κάνα δύο. Πρέπει να συμμετάσχει η νεολαία κοινότητα, η παραπληροφόρηση να η διάκριση, να προστατεύσουμε την υγεία, αναπαραγωγική, η σεξουαλική υγεία των γυναικών. Πρέπει να τι εκπαιδεύσουμε. Πρέπει να τελευταία γενιά αυτή των κοριτσιών που αντιμετωπίζουν τη βία ή αυτή παραβίαση των δικαιωμάτων του μέσω του κρατηρισμού. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνάδελφε Ραφαέλα, έχετε το λόγο. Εκ μέρου του Ρινιού. Καλησπέρα. Θα συνεχίσω Ολλανδικά. 200 εκατομμύρια γυναίκες λοιπόν κάθε μέρα υφίστανται αυτό το μαρτύριο. Φτάνει πια. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε. Είναι άδικο. Στην Ευρώπη επίσης 2.000 γυναίκες καθετός υφίστανται τον κίνδυνο να υποστούν το ίδιο. Δεν μπορεί να σιωπούν. Και ο πόνος είναι κάτι που μένει και πρόκειται για τους συμπολίτε μας. Είναι πολύ σημαντικό να μιλάμε για αυτό το θέμα, αλλά πραγματικά δεν φτάνει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί ώστε να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα και να προστατεύσει τις γυναίκες και τα κορίτσια. Είναι μεγάλο πρόβλημα η βία σε βάρος των γυναικών και ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να φροντίσει αυτή η αδικία να σταματήσει. Ε, ναι, είναι καλό που θέλετε να έχετε μια στρατηγική, αλλά πραγματικά πρέπει να είναι μια σκληρή στρατηγική, μια στρατηγική που να φτάνει σε κυρώσει σε βάρος των υπευθύνων και που θα φροντίσει τέτοιου είδους βία να κοινοποιείται πρώτα απ' όλα. Φροντίστε επίσης και για τις υποδομές σας παρακαλώ και για την χρηματοδότηση, για την πρόληψη πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να φροντίσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες που υπάρχουν και να δώσει η Επιτροπή τη δυνατότητα και στα θύματα για να τα προστατεύσουμε. Φτάνει πια. Πρέπει να έχουμε μια αποτελεσματική στρατηγική. Μια στρατηγική πραγματικά με νύχια και δόντια. Ευχαριστούμε κυρία Κουνκέ εκ μέρους των Πρασίνων. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση συχνά είμαστε πολύ περήφανοι γιατί είμαστε εμείς που υποστηρίζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα παγκοσμίω. Αλλά θα ήταν αστείο να το λέμε αυτό όταν ξέρουμε ότι υπάρχουν τόσες γυναίκες ακόμα και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ακροτηριάζονται κάθε χρόνο. 4.000 ετησίως σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο ε, που είναι αρμόδιο για τέτοια στατιστικά δεδομένα. Και πρέπει να ξέρουμε ότι στην Ευρώπη δεν εκτιμάμε καλά τον κίνδυνο που υπάρχει. Υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος που είναι να θεωρούμε πολιτισμικό φαινόμενο την πρακτική αυτή. Δεν είναι όμως αυτό σωστό. Πρέπει να υποστηρίξουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, να καταπολεμήσουμε τον ρατσισμό και τις πατριαρχικές δομές από όποια κουλτούρα και αν προέρχονται. Ευχαριστούμε. Κυρία Μπίλτ, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε ενώ ένα από τα πρώτα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών κατά του γενετήσιου ακροτηριασμού ανάγεται στο 1952 πάρα πολλές γυναίκες είναι θύματα και τρία εκατομμύρια ε, διατρέχουν τον κίνδυνο να ακροτηριαστούν κάθε χρόνο. Ε, ιδού λοιπόν είναι αποτελεσματικότητα ε, της διεθνούς κοινότητας σε κάτι που συνιστά ωστόσο γενική υπόθεση δικαιολογημένα αναφέρομαι το θλιβερό πεπρωμένο της υποσαχάριας Αφρικής όπου, όπου, στην, ε, όπου υφίσταται τέτοιες πρακτικές σε πολύ μεγάλα ποστά, 35% για παράδειγμα. Ε, αντανάκλαση επίσης της ε, μετανάστευσης ε, είναι το γεγονός ότι πάρα πολλά κορίτσια σε ευρωπαϊκές χώρες υφίστανται αυτές τις πρακτικές. Μία ε, σχετική μελέτη το 2008 το αναγνωρίζει, αναγνωρίζει αυτό το γεγονός. Είδουμε μια, ένα πρώτο βήμα συνειδητοποίησης στο πλαίσιο μιας διαμάχης η οποία παίζεται και στο δικό μας έδαφος. Ε, ε, κυρία που κάθεται στην έδρα 123, λοιπόν, να μην μας δίνει μαθήματα γιατί πρόκειται για τεράστια υποκρισία. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κάθε χρόνο χιλιάδες γυναίκες, νέες γυναίκες είναι θύματα ακροτηριασμού των γενετικών τους οργάνων. Είναι μια πρακτική που είναι βασανιστήριο. Επιβλαβή για τη φυσική και ε, ψυχολογική ακαιρεότητα των γυναικών. Χρειάζονται συγκεκριμένα μέτρα για να τεθεί τέρμα σε αυτή την πληγή. Δεν μπορούμε να δεχτούμε επί της βάσεως παραδόσεων πολιτισμού ή θρησκείας να συνεχίζεται, να εφαρμόζεται αυτή, αυτό το αδίκημα. Είναι θεμελιώδες η διεθνής κοινότητα να έχει μηδενική ανοχή όσον αφορά το θέμα αυτό, αυτού του ακροτηριασμού. Αυτέ τι πράξει που γίνονται σε χιλιάδε. Εκτό τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω κάθε χρόνο και είναι παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου. Η αξιοπρέπεια του ανθρώπου πλήττεται. Η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι αξίε θεμελιώδη του ευρωπαϊκού εγχειρήματο. και ήδη προβλέπεται ω ποινικό αδίκημα σε όλα τα κράτη-μέλη. Όμω σύμφωνα αν βάλουμε το δάκτυλο επί του τύπου των ύλων, βλέπουμε ότι είναι πολύ λίγε καταδίκε στα δικαστήρια. Θα πρέπει να στατεύουν τα κράτη-μέλη καλύτερα τα κορίτσια και τι γυναίκε. Είναι θεμελιώδε αυτοί που διαπράττουν αυτά τα δικήματα εντό και εκτό ενώσεω να τιμωρούνται, να δικάζονται και να τιμωρούνται. Εμπλεκόμενοι και η κοινότητα μέσω ευαισθητοποίησεω ε, για αυτή τη μάστιγα. Έτσι θα πετύχουμε μόνο τον στόχο του ΟΗΕ τη εκρίζωσης της πλήρους εκρίζωσης της πρακτικής μέχρι το 2030. Ελπίζω ότι αυτή θα είναι και μια προτεραιότητα της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να είναι στην πρώτη γραμμή σε αυτή την μάχη. Ευχαριστώ πολύ. Συνάδελφε Λαϊτάου Μάρκες από Σοσιαλιστές και Δημοκράτες έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, ε, κυρία Υπουργέ. Η έγκριση μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για την καταπολέμηση του γενετικού κριτηριασμού των γυναικών είναι κάτι θεμελιώδες. Πρέπει να καταπολεμηθεί σε όλο τον κόσμο. Οι κοινωνικές συνθήκες, οι θρησκευτικέ παραδόσεις, τα στερεότυπα που συνδέονται με τη γυναικεία σεξουαλικότητα δεν πρέπει να συνεχίζουν να είναι κίνητρο για να δημιουργούν ανεπανόρθωτη ζημιά στα σώματα των γυναικών και των νέων κοριτσιών δυστυχώς υπάρχουν ελάχιστα σίγουρα στοιχεία όσον αφορά αυτή τη μάστιγα που ήδη θα έπρεπε να είχε εξαφανιστεί τον 21ο αιώνα. Γνωρίζουμε ότι περίπου 200 εκατομμύρια θύματα έχουμε στον κόσμο. 50 εκατομμύρια από αυτά τα θύματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό έχουμε τρει σημαντικέ πτυχέ. Καταρχά, τα κράτη-μέλη πρέπει να συλλέγουν περισσότερα στοιχεία για το φαινόμενο στι διάφορε χώρε και να συμμετέχουν περισσότερο οι επαγγελματίε του τομέα τη υγεία για την καταπολέμηση στην αποτελεσματική του φαινομένου. Δεύτερον, θα πρέπει να υποστηρίξουμε καινοτόμε λύσει που θα εδράζονται επί τεχνολογία, όπω παραδείγματο χάρη το, η ICOT, ε, η εφαρμογή αυτή που χρησιμοποιείται στην Κένια, που δημιουργήθηκε από αυτή την ομάδα των νέων γυναικών που συναντήσαμε και ελπίζουμε να μπορέσουμε εκ νέου να τις προσκαλέσουμε βλέποντας ότι βραβεύτηκαν σε αυτή τη μάχη τους. Θα πρέπει να ακυρωθεί και η σύμβαση της Κωνσταντινούπολη που προβλέπει αυτό ότι ο κριτηριασμός είναι ποινικό αδίκημα. Δεν, θα παραμένουμε, δεν πρέπει να παραμείνουμε αδρανείς όσο υπάρχει ακόμα έστω και μια γυναίκα που είναι θύμα αυτού του κριτηρισμού. Ευχαριστώ συνάδελφε Άντρουλε για το ID. Έχετε το λόγο. 500.000 γυναίκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν θύματα γενετικού ακροτηριασμού και κάθε χρόνο 180.000 περισσότερε θα αντιμετωπίσουν αυτό το κίνδυνο. Έχουμε από το ίντερνετ του Κοινοβουλίου και έχουμε διάφορα σχόλια. Γενετικό ακροτηριασμό των γυναικών ακόμα ακολουθείται σε διάφορε αφρικανικέ χώρε, στην Ασία και στη Μέση Ανατολή. Λοιπόν, με μία λέξη, αυτή η φρικόδης πρακτική ε, δεν έχει μόνο βάση ε, ευρωπαϊκή, δεν έχει βάση ευρωπαϊκή, αλλά σκείται και στην Ήπειρό μας. Θα πρέπει να κάνουμε τα αναγκαία στα του οίκου μα πριν κινηθούμε προ τα έξι. Γιατί φτάσαμε μέχρι εκεί. Είναι, έχουμε, εισάγουμε ανθρώπινα όντα και τι πρακτικές τους, ακόμα και τι πιο απάνθρωπες στο βαθμό που δεχόμαστε μια μετανάστευση αναρχική, δίνουμε ελεύθερο, δεύτερη είσοδο στη βία. Εδώ στη Γαλλία οι γυναίκες, οι ενήλικε που έχουν ακροτηριαστεί από 62.000 το 2000 έφτασαν 184.355 την αρχή τη δεκαετία μα. Λοιπόν, ε, ε, είναι βία που διαπράτεται στο σώμα τους και βία κατά των γυναικών. Ανοίξουμε τα μάτια. Δεν μπορούμε να λεγόμαστε ότι είμαστε φεμινίστες και να επικροτούμε χιλιάδε μεταναστών που περιφρονούν τη γυναίκα ή καμιά φορά την κακομεταχειρίζονται ή βιοπραγούν εναντίον της. Η, η Ευρώπη θα μπορούσε να περιναυτεί ότι δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιεί, χρησιμοποιεί σκοτεινέ πρακτικέ να βλάπτει τα κορίτσια σα. Αλλά προτιμάμε, βλέπετε, να δεχόμαστε τα πάντα λόγω ορθή πολιτική πρακτική, politically correct. Λοιπόν, ε, ενώ με το σεβασμό τη γυναίκα, θα πρέπει να αποκαταστήσουμε τι ευρωπαϊκέ αρχέ ε, στο καταστατικό μα. Ευχαριστώ πολύ. Συνάδελφε Πόσπισιλ, έχετε το λόγο εκ μέρου του ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, σας άκουσα με πάρα πολύ προσοχή και ενδιαφέρον για την πρωτοβουλία σας που σίγουρα θα τύχει τη στήριξη του Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίου. Και χαίρομαι που οι περισσότεροι ομιλητές βλέπουν τον κίνδυνο αυτό πάρα πολύ σοβαρά, τον κίνδυνο σε βάρος των γυναικών. Και εγώ βλέπω δύο πτυχές. Πρώτον, υπάρχει η βία και που υπάρχει και εδώ στην Ευρώπη. Και δεύτερον, η βία σε άλλα σημεία του κόσμου. Χρειαζόμαστε μέσα και για τις δύο περιπτώσεις διαφορετικά όμως. Τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρέπει να επικεντρωθούν στην βία, στην Ευρώπη επίσης, γιατί είναι πραγματικά τροπή να υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες ή και εκατοντάδες χιλιάδες περιπτώσεις τέτοιου ακροτηριασμού στην ε, Ευρώπη πρέπει να πούμε στους ανθρώπους αυτούς ότι κοιτάξτε εσείς έρχεστε στην Ευρώπη, ζείτε στην Ευρώπη, πρέπει να σεβαστείτε τις ευρωπαϊκές αξίες και πρόκειται εδώ για ανθρώπινα δικαιώματα και ισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Πολλά λοιπόν έχουμε να κάνουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Οι αρχέ συμμόρφωση επίση πρέπει να ασχοληθούν περισσότερο. Εάν κάποιο προβαίνει σε αυτό το έγκλημα, πρέπει να διώκεται και να καταλήγει στη δικαιοσύνη. Χρειάζεται και συνεργασία μεταξύ των χωρών μελών, κάτι που δεν είχαμε μέχρι τώρα. Ξέρουμε ότι έχουμε χιλιάδε δεκάδε. χιλιάδε τέτοιες περιπτώσεις, αλλά πραγματικά, ρεαλιστικά, πόσοι από αυτού κατέληξαν στη δικαιοσύνη. Πόσοι καταδικάστηκαν. Κάτι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Συγχρόνω πρέπει να δουλέψουμε και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πάρει περισσότερο χρόνο σίγουρα, αλλά καταρχήν να δουλέψουμε πάνω σε αυτό το πρόβλημα στην Ευρώπη. Το χρωστάμε αυτό, το οφείλουμε σε όσους έρχονται εδώ και πρέπει να προστατεύουμε τα δικαιώματά τους. Ευχαριστούμε. Τάξη, σοσιαλδημοκράτες. Ευχαριστώ. Φανταστείτε, είσαστε 8 χρονών κορίτσι.